Ε, εδώ που είναι το μηχάνημα κάθισε ο γραμματέας και ο πρόεδρος της Επιτροπής χαίρεται διότι βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο. Όλα είναι συμβολισμοί των συσχετισμών δυνάμεων εδώ στο Κοινοβούλιο. Αμέσως περνάμε στην ψηφοφορία. Ε, η μερίσια διάταξη προβλέπει και μια σύντομη συζήτηση με τον εκπρόσωπό μας στην Μιανμάρ. Ε, τα έχουμε συμφωνήσει όλα αυτά και περνάμε στην ψηφοφορία. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Ο εισηγητής μας είναι ο συνάδελφος Αλαφράνκα. Θέλετε να λάβετε το λόγο κύριε Σαλαφράγκα. Όχι. Ωραία. Οπότε προχωρούμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ε, προφορική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ε, 50-78 υπέρ κατά αποχές ε, 5.000 ε, κατά δεκτή. 5.001 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 50.79 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50.80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 51.24 υπέρ, κατά αποχές δεκτό. 5.002 υπέρ, κατά αποχές δεκτό, 50.81 υπέρ, 5081 μεχρι 5087 όλες μαζί αν συμφωνείτε. Ναι, συμφωνεί και ο συντάκτης υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 5.003 ε, υπέρ, κατά. Ξαναψηφίζουμε. 5.003 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 50.89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50.04 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 50.90 υπέρ 50-90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-05 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51-28 υπέρ κατά Απορρίφθηκε. Προφορική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 50-06 περα κατα Κατά αποχές δεκτή. 50-93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50-07 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 50-92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-08 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50-94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-09 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50-10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50-11 υπέρ κατά αποχές δεκτή Προφορική τροπολογία 7. Υπέρ. Πρόεδρε, ζητώ το λόγο για την τροπολογία 51-30 μετά από την 7. Τότε θέλω το λόγο, παρακαλώ. Προφορική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Και τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε κάποιες αμφιβολίες για την τροπολογία αυτή της κυρίας Γιατεμάκη. Για να υπάρχει συνοχή δηλαδή με την περσινή μας ψηφοφορία, θα την ψηφίσουμε αν και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για τη βιωσιμότητα μιας γραμμής για τον καθέναν από τους ειδικού απεσταλμένους. Γι' αυτό θέλω να αλλάξει η ψηφοφορία της ομάδας μου και να πω στην ομάδα μου ότι θα υπερψηφίσουμε αυτή τη φορά. 51-30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ. Κατά πίπτη. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, προφορική τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 37 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 95 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ποιος είναι υπέρ της 112, ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 112. Πέρα της ψηφοφορίας. 47. Όχι, όχι. απορρίφθηκε 21 κατά 21 ε, προς 21 99 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 114 υπέρ. Κατά έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Γιατί είναι 25 προς 24. 25 είναι τα υπέρ. Εκατόν ένα, προχωρούμε. Πρόεδρε, δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου. Ε, απέχω, να ξέρετε. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Ψήφισα αποχή. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα με τις ε, τρεις αποχές. Αντί για Προχωρούμε. Μπορείτε να πάτε στην ε, διπλανή θέση. Ε, υπάρχει πρόβλημα. 101. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά δεκτή έλεγχος πρέπει να είστε καλύτερα, να φέρεστε καλύτερα, να είστε πιο ευγενικοί προς τους συμπατριώτες σας, κυρία Μουνίθ. Πέρας. 25 προς 24 δεκτή. 129 υπέρ. Συγγνώμη, αλλά ε, ε, δείχνει 24-24. Είναι και η δική μου η ψήφος. Συν τη δική μου ψήφο, λέει ο πρόεδρος, γι' αυτό είναι 25 που δεν έχω το μηχάνημα μπροστά μου. 129 υπέρ. Κατά. θα πρέπει εφόσον δεν λειτουργεί το μηχάνημα να ε, αλλάξει θέση ο συνάδελφος ή να φωνάξει τον τεχνικό. 129 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, έλεγχος. Πέρας. Απερίφθη. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Πέρας. Απερίφθη με διαφορά μιας ψήφου 23 υπέρ 24 κατά 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 118 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απερίφθη με, την ίδια, με τον ίδιο συσχετισμό όπως και πριν. 50-21 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 105 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 58 καταπίπτει. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 126 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Παρακαλώ, κυρία Μουνίθη. Ζητήσαμε για την για την 119 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία. Ist geschlossen. Πέρας. Απερίφθη. 22 υπέρ 24. κατά. Τώρα που είχαμε φτάσει... Και την 127 ψηφίσαμε. 121. Εκεί φτάσαμε. 121 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 με την 9 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, προφορική τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 75 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 30 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 3 ε, υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 34 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ε, ναι, ναι, το ίδιο είναι το αποτέλεσμα, δεν έπρεπε να ψηφίσουμε, είχε καταπέσει. 120 ε, υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 77 υπέρ. Α, και αυτή καταπίπτει. Ωραία. Και αυτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά έλεγχος 70 άρχεται η ψηφοφορία 25 προς 27. Όχι, 24 προς 28. Απερίφθη. Η 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Äh, Πάμε λοιπόν τώρα στη γνωμοδότησή μας για τον ε, προϋπολογισμό και η συγητής είναι και πάλι ο συνάδελφος κύριος ε, Σαλαφράνκα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει από αυτού. Πάμε λοιπόν στην ψηφορία. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Εδώ πρόκειται για την ψηφοφορία για ένα μόνο κομμάτι αυτής της πρότασης. Υπέρ παρακαλώ. Τέσσερα. Ψηφίζουμε για την τέσσερα με την τροποποιημένη της μορφή. Υπέρ παρακαλώ για την 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται εδώ. Πρόκειται για προγράμματα της ε, πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μήπως εννοείται ότι το πρώην Ανατολική Γερμανία ε, σημαίνει κατ' ουσίαν αφοπλισμός deutsche Demokratische Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά αποχές για την 8 παρακαλώ. Για άλλη μια φορά 8. Υπέρ Ποιος είναι υπέρ της 8. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. για την 12 ψηφίζουμε μόνο το κομμάτι που λέει Especially Severe External Action. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Επίσης... Ε, Ψηφίζουμε για ένα συγκεκριμένο τμήμα αυτής της πρότασης. Υπέρ της 13 κατά αποχές εγκρίνεται. 14 κατά καταπίπτει ή 15 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 η 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 32 υπέρ, καταπίπτει, καταπίπτει η 32, 33 και 34 υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπορική προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, υπέρ παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η γνωμοδοτήση 48-5 και μία εποχή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στη γνωμοδότηση του συναδέλφου Κατσίν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κατσίν θέλει να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Τροπολογία υπερθμών 1 παρακαλώ, με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η τέσσερα Έχει αποσυρθεί. Η 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον εγκρίνεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε με αποτέλεσμα 32 υπέρ, 21 κατά. Η 7 σε δύο τμήματα, το δεύτερο τμήμα βέβαια έχει αποσυρθεί, άρα ψηφίζουμε μόνο για το πρώτο, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 11 υπέρ, κατά εγκρίνεται, η 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της, ε, των, της γνωμοδότησης, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, έκλεισε η ψηφοφορία, έχει κλείσει η ψηφοφορία. 53 προς 1, ε, καλύτερα να πούμε 54. 54 ψήφισαν υπέρ. Σας ευχαριστώ θερμά.